Good morning, everyone. First of all, I would like to wish you a happy and successful new year. Καλή χρονιά. Ε, εύχομαι σε όλους σας. Αρχίζουμε αμέσως με το σημείο 1 της ημερήσιας διάταξης, έγκριση αυτής. Νομίζω όλα είναι εντάξει. Δεύτερον, έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 9ης ε, Δεκεμβρίου, 5ης και Δευτέρας Δεκεμβρίου. Είναι εντάξει. Και έχουμε και ένα επιπλέον σημείο, το οποίο είναι η διαβούλευση βάσει του άρθρου 70 του κανονισμού κτλ. Τρία θέματα έχουμε βάσει το άρθρο 70, επί των οποίων επετεύχθη συμφωνία στο Συμβούλιο στα τέλη της Λιθουανικής Προεδρίας. Και αυτά είναι η οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίαση των τραπεζών, για ε, την κατάχρηση της αγοράς και για την εγγύηση των καταθέσεων. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, για τις τράπεζες έγινε ένα συμβιβασμός με τη Λιθουανική Προεδρία στις 11 Δεκεμβρίου στον τριμερή διάλογο του 2013 και τεχνικά ολοκληρώθηκαν όλα αυτά ε, νωρίς τα ξημερώματα της 18ης. Το Κορεπέρ το ενέκρινε αυτό στις 20 Δεκεμβρίου στη συνέχεια και η επιστολή που το επιβεβαιώνει ελήφθη ε, την ίδια μέρα το απόγευμα. Καλύπτεται από το νέο άρθρο 70 του κανονισμού αυτό και καλούμεθα να ψηφίσουμε τυπικά και επίσημα. Ε, υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, ετοιμάζεται λοιπόν για έγκριση σε πρώτη ανάγνωση στην Ολομέλεια. Sorry for ε, Συγγνώμη για τον καφέ. Λοιπόν, ε, σε ό,τι αφορά την οδηγία για το σύστημα εγγύηση καταθέσεων, 17 Δεκεμβρίου ήταν ο τριμερής διάλογος πάλι. Η τεχνική εργασία ολοκληρώθηκε στις 19-12 του 2013. Όπως ε, και με την οδηγία για τις τράπεζες ε, η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων το ενέκρινε στις 20 Δεκεμβρίου. Το Κοινοβούλιο έχει ολοκληρώσει εδώ την πρώτη του ανάγνωση και σε περίπτωση που εγκριθεί ε, το θέμα θα γίνει ε, ε, νωρίς η δεύτερη ανάγνωση και θα υποβάλουμε την άποψή μας στο Συμβούλιο. Δεν έχουμε λάβει επιστολή από το ΚΟΡΕΠΕΡ. Αν συμφωνεί το Συμβούλιο σε πρώτη ανάγνωση, προτείνει ο Πρόεδρος να εγκριθεί το ίδιο κείμενο σε δεύτερη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο. Θα ψηφίσουμε λοιπόν διανατάσσεως χειρός υπέρ και για αυτό το θέμα κατά αποχές. Η Πρόεδρος λοιπόν θα απευθύνει επιστολή στο Συμβούλιο σύμφωνα με τα όσα σας είπα. Ε, ε, σας είπα. Τι σημαίνει αυτό για το χρονοδιάγραμμα πλέον για την Ολομέλεια. Μόνο τον Απρίλιο μπορεί να εγκριθεί. Τώρα για την εξυγίαση των τραπεζών, την αντίστοιχη οδηγία, έχει προγραμματιστεί για τη δεύτερη ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Ταυτόχρονα συνδέονται, γνωρίζετε σημαντικά οι δύο αυτές εκθέσεις και ο μηχανισμός ε, ε, δεν χρειάζεται να το αποφασίσουμε τώρα αυτό, θα το έχουμε υπόψη μας. Οι εισηγητές θέλουν να πούν τίποτα για τις εκθέσεις τους αυτές. Όχι, καλώς. Λοιπόν, προχωρούμε. Διαβούλευση για την οδηγία για τις ποινικέ κυρώσεις για την ε, κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών και αγοράς. Σύμφωνα ε, πάντα με το άρθρο 70 θα πρέπει να αποφανθεί η Επιτροπή μας ε, επιτεύχθη συμφωνία για όλα τα θέματα μετά από το πολιτικό τριμερή διάλογο στις 10 Δεκεμβρίου και στις 17. Το τελευταίο τελικό κείμενο κυκλοφόρησε στις 19 για τους κοιόδης συγητές και τις πολιτικές ομάδες, ενώ στις 20 του το ενέκρινε η Κορεπέρ και έστειλε και επιστολή την ίδια μέρα. Ε, ε, η κυρία Μακάρθη θέλει να πει τίποτα γι' αυτό. Πολύ σύντομα. Προφανώ θέλω να ευχαριστήσω του σκιώδη ηγητέ που έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και ήμασταν πραγματικά ενωμένοι, στοιχημένοι και πολύ σκληρή ήταν η μάχη και η συμφωνία τελικά με το Συμβούλιο. Εξαιρετικοί πάντα οι υπάλληλοι που του παραμελούμε καμιά φορά και του ε, λησμονούμε ε, για να ρυθμίσουν τα τεχνικά. Θα ήθελα να πω ευθύ εξ αρχή το εξή, μια που πάμε και σε ευρωεκλογέ και ποια είναι τα θέματα που μα ενδιαφέρουν μα ω Επιτροπή και ω Κοινοβούλιο και τι αποτελέσματα προσφέρουμε. Είναι πολύ σημαντικό που έχουμε τώρα ποινικέ κυρώσει παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση για κατάχρηση των αγορών και έχουμε και μια ελάχιστη ποινή φυλάκιση, αν μη τι άλλο. Για την Επιτροπή Ελευθεριών ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Το Συμβούλιο ούτε να τα ακούσει Είπαμε εμείς θα ορίσουμε ποιες θα είναι οι ελάχιστες κυρώσει, αλλά τελικά ε, επιτύχαμε την, μια ελάχιστη ποινή φυλάξη που είναι τέσσερα έτη ε, για την ε, ε, εσωτερική προφόρηση και ε, για την αποκάλυψη διετία. Έχουμε την χρηματοπιστωτική κρίση και τα διάφορα νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται εκεί θα λογοδοτούν και θα ε, υφίστανται και ποινικέ κυρώσει. Θα είναι και ποινικά υπεύθυνοι. Για πρώτη φορά εταιρείε δηλαδή παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ε, λογοδοτούν. Υπήρχε αυτό σε μερικά κράτη-μέλη, όχι σε όλα. Υπάρχει και το θέμα της βαριάς αμέλειας για πρώτη φορά, σοβαρής, αυτό το recklessness στα αγγλικά ε, αν υπάρχει λοιπόν βαριά σοβαρή αμέλεια, ε, έστω και αποσία δόλου μπορεί να στοιχειοθετηθεί ποινική ευθύνη. Αυτά. Και επίση θα δημοσιεύονται οι κυρώσεις αυτές και μπορείτε όλοι να το διατρανώσετε αυτό στην προεκλογική εκστρατεία για να διαφημίσουμε τι έκανε το Κοινοβούλιο προς όφελος των Ευρωπαϊκών. Ευχαριστώ και πάλι τους συναδέλφους για την υποστήριξή τους. Ευχαριστώ πολύ, Αρλίν. Αν δεν διαφωνεί η Επιτροπή, θα θεωρήσω ότι έχουμε καταλήξει ε, σε συμφωνία για το κείμενο το συμβαστικό που θα καταδεχθεί στην Ολομέλεια. Πότε το Φλεβάρι, την πρώτη σύνοδο. Ωραία, ευχαριστώ. Θα ήθελα να υποβάλω ένα ε, ερώτημα ως προς τις ε, ποινικές κυρώσεις. Ξέρουμε ότι δεν είναι πολύ εύκολες. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τις δυνατότητες ως προς τις διοικητικές κυρώσεις που είναι και πιο εύκολες. Τι δυνατότητες υπάρχουν. Συμφωνήσαμε τον Ιούλιο από αυτόν. Οι ποινικέ ήταν το δεύτερο μέρος της οδηγίας κάτι το οποίο ήταν πιο δύσκολο στη διαπραγμάτευση και επειδή έπρεπε να το δούμε μαζί με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, επειδή υπήρχε ενισχυμένη συνεργασία, το κάναμε, δηλαδή τις ε, καταχρήσεις ως προς την αγορά της ε, διακινήσεις στην αγορά. Γι' αυτό θα σας αποστείλω ε, ένα κείμενο για να δείτε τι έχουμε επιτύχει ως προς τις διοικητικές ε, κυρώσεις. Το κάναμε τον Ιούλιο, θα το ξανακάμε το Φεβρουάριο για να έχουμε ένα ε, πλήρες πακέτο. Σαν Πολ κάτι άλλο, όχι. Επόμενο θέμα. Η Επιτροπή. delegated act under CRR. The dele the dele σε σχέση με τις ε, κατεξιοδότηση πράξεις, στις 6 Ιανουαρίου αποφασίσαμε και ως προς την Ως προς την οδηγία για τις κεφαλιακές απαιτήσεις προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να αποτιμήσουμε και να προσαρμόσουμε την κατάσταση δυνάμει του άρθρου 110. Το Κοινοβούλιο έχει ένα μήνα μέχρι τις 20 Ιανουαρίου για να εγκρίνει τις κατεξιοδότηση πράξεις πριν, ε, και, πριν, και επειδή ακριβώς είχαμε διακοπές, είχαμε τις διακοπές, ήταν πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να ευθυγραμμιστούμε με τον ένα μήνα. Εξ ονόματος της ΕΚΟΝ λοιπόν θα ζητήσω παράταση της διαδικασίας ελέγχου κατά ένα μήνα όπως προβλέπεται από το άρθρο 463 του Κανονισμού για την Κεφαλαιακή Επάρκεια. Σε σχέση με το MIFID ΜΥΦΙΝ, συγγνώμη, στις 18 Δεκεμβρίου προβλέψαμε ένα διάλογο για να δούμε και τα παράγωγα και την πρόσβαση στην αγορά το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού και της κυρώσης Επίσης έχει επιτελεστεί πρόοδος και είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία, αλλά υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα τα οποία χρήζουν περαιτέρω συζήτησης. Για τις 14 Ιανουαρίου προβλέπεται τριμερής διάλογος σε σχέση με τα αποθετήρια ε, κινητών αξιών. Έχουμε, είχαμε προβλέψει τριμερή διάλογο στις 18 Δεκεμβρίου και λάβαμε υπόψη και τα βοηθητικά μέσα για την ε, αντιμετώπιση των ε, ζητημάτων που αφορούν την Τραπεζική Ένωση. Προβλέπουμε τριμερή διάλογο και θα ακολουθήσουμε την ε, γνωστή, την προβλεπόμενη οδό. Σε σχέση με το μηχανισμό εξυγίανσης τραπεζών στις 13 Ιανουαρίου θα αποφανθούμε επί του θέματος. Λοιπόν, τώρα θα ασχοληθούμε με τα θέματα 4, 5 και 6, δηλαδή την απαλλαγή 2012 της Ευρωπαϊκής ε, Αρχής Τραπεζών, την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Ο Αντολίν Σάντσες Πρεζέδο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρο. Εντάχει θα παρουσιάσω το όλο ζήτημα, αυτή τη γνωμοδότηση για την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού σε σχέση με την απαλλαγή του 2012 για την Ευρωπαϊκή Αρχή ε, Τραπεζών την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Η απαλλαγή αφορά το 2012. Είναι η δεύτερη έκθεση που συντάσσεται για αυτό το θέμα. Ο Μπερνάρ Λάγκεν είχε συντάξει την πρώτη και λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της στιγμής. πρόκειται για μια διαδικασία πληρέστερη από την πρώτη μέσα στα πλαίσια της απαλλαγής σε σχέση με τη λειτουργία των αρχών. Όπως ξέρετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο στην εκπόνηση του ζητήματος καθώς και τις ευθύνες που φέρει κάθε αρχή. Λαμβάνοντας υπόψη και την εισήγηση του ελεγκτικού συνεδρίου, γιατί ξέρετε ότι έχει συντάξει τρεις εκθέσεις για κάθε μία αρχή ξεχωριστά, ως προς τους ετήσιους λογαριασμούς των τριών αυτών αρχών και την, το οικονομική την οικονομική κατάσταση των αρχών. Οι λογαριασμοί πληρούν όλους τους όρους που προϋποτίθενται και αυτό είναι και το σημείο εκκίνησης. Υπάρχουν ε, ορισμένα ζητήματα στα οποία επέμεινε το ελεγκτικό συνέδριο στην πρώτη αυτή έκθεση και ε, χρειάζονται σχόλια και μέσα που θα πρέπει να προωθηθούν και το ίδιο το ελεγκτικό συνέδριο αξιολόγησε την κατάσταση όπως όφιλε και με βάση την προηγούμενη έκθεση. Γι' αυτό προσπάθησα να φτάσω σε έναν απολογισμό με βάση τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Υπάρχουν όμως ζητήματα τα οποία θα πρέπει να προωθήσουμε περαιτέρω. Για την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, για παράδειγμα, το 12 είχαμε 20 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμό, 8 εκατομμύρια για κοινοτικά ζητήματα και 12 αφορούν τα κράτη-μέλη. Και βεβαίως υπάρχει ένα μικρότερο κονδύλι για τους παρατηρητές. Αυτό που έχει σημασία είναι πώς, ελέγχονται, πώς ελέγχεται η χρήση αυτών των κονδυλίων και γι' αυτό θα μπορούσαμε να προβούμε σε ορισμένες τροποποιήσεις. Το ελεγκτικό συνέδριο έκρινε ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η διαφάνεια μέσα στα πλαίσια της πρόληψης, πρόσληψης προσωπικού και έλεγχος των συστημάτων πληροφορικής. Παράλληλα, τόνισε ότι οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να ε, στηρίξουν την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών υπάρχουν 15 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια για την, ε, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε μια αύξηση 50% το 2012. θα πρέπει να προβούμε σε διορθωτικές ε, πράξεις σε σχέση με, τα, με τις ε, κινητές αξίες και μέσα στα πλαίσια της, ε, των προσλήψεων θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Επέμενε, επέμεινε από αυτού το ελεγκτικό συνέδριο και θεωρώ ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ως προς την Ευρωπαϊκή Αρχή ε, Κινητών Αξιών και ε, Αγορών, 20 εκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός, όπου το κοινοτικό σκέλος είναι 7 εκατομμύρια, αφορά 7 εκατομμύρια Και εδώ χρειάζονται διορθωτικές πράξεις, μερικές έχουν ήδη προωθηθεί και θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, η αξιολόγηση των λογιστικών συστημάτων και η αποτίμησή τους ε, η βελτίωση των συστημάτων πληροφορικής και βελτίωση του συστήματος πρόσληψης προσωπικού. Πέρα από αυτά, υπάρχουν δύο άλλα ζητήματα. Ποια θα είναι η δημοσιονομική εξέλιξη εάν λάβουμε υπόψη ότι πρόκειται για αρχές που δεν έχουν οριμάσει, που τώρα έχουν θεσπιστεί και συσταθεί και ο προϋπολογισμός του 2014 ορίζει τον, τον περιορισμό και τα όρια των προϋπολογισμών αυτών των τριών αρχών. Για το 2015 θα πρέπει να υπάρχουν, να προβλεφθούν περισσότερα κονδύλια. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ιδιαίτερα για την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και Κινητών Αξιών. Επίσης, το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα υποστήριξε την αυτονομία αυτών των αρχών μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού και τώρα που, θα, ε, που θεσπίστηκε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Εποπτείας θα πρέπει να δούμε πώς θα, είναι, πώς θα έχει και η εξέλιξη αυτών των τριών αρχών ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια του ενιαίου μηχανισμού εποπτείας. Αυτά είναι τα στοιχεία που θα ήθελα να σας υποβάλω και θα ήθελα να ε, μου προβάλετε υποδείξεις για να φτάσουμε σε ένα πολύ καλό τελικό αποτέλεσμα και σε συμφωνία. Ευχαριστούμε πολύ Αντολίν. Εξ ονόματος του ΕΛΚ δίνω το λόγο στην κυρία Γκάλπες. Ε, Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Σάντσες Πρεσέτο για την διεξοδογικότατη παρουσίαση της έκθεσής του. Ε, είναι εξαιρετικά τεχνικής φύσεως το θέμα Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα αυτές οι αρχές και άρα θα πρέπει, ε, οφείλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το ζήτημα. Ε, το είχαν ανατεθεί ε, καθήκοντα, εξουσίες, αρμοδιότητες σε αυτές τις αρχές που βρίσκονται στον πύρινα των δραστηριοτήτων της δικής μας Επιτροπής. Συμφωνώ με τα πορίσματα της έκθεσης ε, του ελεγκτικού συνεδρίου και τα διορθωτικά μέτρα που εισηγείται το, συνέδριο, το ε, ελεγκτικό συνέδριο ως προς ε, τη διαφάνεια κατά την διαδικασία επιλογής, παραδείγματος χάρη τη μείωση του κόστους, υιοθέτηση νέων μοντέλων διαχειριστικών και ούτω καθεξής. Αυτές οι εποπτικές αρχές Όλες αυτές οι αρχές έδωσαν ε, τάχιστα απαντήσεις ε, στις παρατηρήσεις ε, της έκθεσης του ελεγκτικού συνεδρίου και έχουν ήδη δρομολογηθεί, έχει δρομολογηθεί εφαρμογή των διορθωτικών μέτρων. Πρέπει επίσης να εξετάσουμε τη δημοσιονομική πτυχή των πορισμάτων. Ενδέχεται να μην ήταν τελείως ο δημοσιονομικός σχεδιασμός, όμως αυτό θα είναι και αναμενόμενο, διότι είναι νεότευτοι οι οργανισμοί, οι αρχές αυτές. Ευελπιστούμε λοιπόν να βελτιωθεί ο δημοσιονομικός σχεδιασμός στο μέλλον. Θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο επ' αυτό. Ίσως να μην χρειαστεί ε, ξεχωριστή γραμμή στον προϋπολογισμό. Ίσως ένα ε, επιμέρους τμήμα γραμμής του προϋπολογισμού θα αρκούσε ούτως ώστε να ε, ε, διευκολυνθεί και το δικό μας έργο. Για την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών θα συμφωνήσω και πάλι με το ελεγκτικό συνέδριο. Εφόσον μιλάμε για την εποπτική αρχή, είναι ρηψοκίνδυνο το σύστημα πληροφορικής να ανατεθεί εξωτερικά σε τρίτο μέρος, κυρίως δε επειδή αυτό συνεπάγεται ένα υψηλότερο κόστος. Η διαδικασία προσλήψεων για την Ευρωπαϊκή Αρχή ε, Τραπεζών αλλά και για την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών ε, Αξιών είναι ένα ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί ε, πιο εξανυχιστικά, διότι προς το παρόν δεν μπορούμε παρά να τονίσουμε ε, πόσο υποδειγματική ήταν η συνεργασία με αυτές τις αρχές, όμως δεν έχουμε απευθύνει επαρκείς κριτικές για αυτό το ζήτημα των προσλήψεων. Για τους ανθρώπινους πόρους γενικότερα θα έλεγα ε, πως επιδέχεται η λειτουργία των αρχών βελτιώσεις Νομίζω ότι συγκεκριμένα για τις προσλήψεις, ε, κυρίως επειδή βρισκόμαστε σε πρώιμο στάδιο, θα ήταν πιο λογικό να ανακατανύμουμε τα καθήκοντα παρά να ε, προσφύγουμε σε αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων, προς το παρόν τουλάχιστον. Ταυτόχρονα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τους απαιτούμενους ε, δημοσιονομικούς πόρους ε, για τις αρχές αυτές, ώστε να λειτουργήσουν εύρυθμα. Εν γέννη θεωρώ ότι ε, δεν είναι ιδιαίτερα προβληματική η κατάσταση και ότι θα καταφέρουμε εύκολα να καταλήξουμε συμβαστικές προτάσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκάλ Πέλτς, εξ ονόματος των φιλελευθέρων. Το λόγο έχει η κυρία Γιάνσεν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Σάντσις ε, Πρεσέντο για τις ε, εξηγήσεις που μας έδωσε για τις τρεις ε, ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές. Συμφωνώ απολύτως μαζί του. Νομίζω δε ότι ε, κατάφερε να τονίσει τα πλέον σημαντικά ε, στοιχεία ε, ως προς τη λειτουργία αυτών των τριών εποπτικών αρχών. Οι τροπολογίες μου είναι μάλλον καλοπιστικές, δηλαδή θέλω να διευκρινίσω κάποια σημεία και όχι να τροποποιήσω το περιεχόμενο της έκθεσής του. Στο σημείο 7 βλέπουμε την ουσία ε, των διευκρινήσεων που μας δίνει ο κύριος Σάντσες Πρεσέντο, διότι εκεί μιλάμε για την χρηματοδότηση ε, που προέρχεται από τις ε, εθνικές αρχές και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα είναι η ανεξαρτησία αυτών των οργανισμών. Γι' αυτό το λόγο έχει ε, σημασία ε, ο ρόλος μας να κατοχυρώσουμε ένα εν μέρη τουλάχιστον ε, προϋπολογισμό εν μέρη, μία εν μέρη χρηματοδότηση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργία αυτών των εποπτικών αρχών και να θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε επίσης σε ποιος είναι ο ρόλος των Εθνικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ε, μην ξεχνάμε ότι κάποια κράτη-μέλη δεν θα τηρήσουν τα υπεσχημένα για τη χρηματοδότηση. Αυτό όμως ε, θα αποτελέσει ε, κόλλημα για τη λειτουργία των εποπτικών αρχών. Ή εάν καταβληθούν υπερβάλλοντα ποσά θα πρέπει να ανακτηθούν στη συνέχεια από τις εποπτικές αρχές. Πώς λοιπόν θα γίνει η ανακατανομή κυρίως σε ε, επίπεδο τριμήνου ανάμεσα σε 28 κράτη-μέλη. Ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Στη συνέχεια υπάρχουν 28 διαφορετικοί δημοσιονομικοί κανονισμοί, 28 διαφορετικοί εθνικοί ε, δημοσιονομικοί οργανισμοί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ο συντονισμός και παρότι αυτό μπορεί να μας εξασφαλίσει τα, τα, τα χρήματα που χρειαζόμαστε, το ρευστό ας το πω έτσι, δεν νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος ε, ε, για να προχωρήσουμε. Τώρα, Πρόεδρε, και εγώ είμαι στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών και όπως ξέρετε ε, ασχολούμαστε τώρα με τον προϋπολογισμό 2014 και αγωνιστήκαμε για να εξασφαλίσουμε τα απαιτούμενα κονδύλια για τις τρεις εποπτικές αρχές. Λοιπόν, θα χρειαστεί να φροντίσουμε για τη μελλοντική λειτουργία των εποπτικών αρχών, ούτως ώστε να αποκτήσουν εν τέλει ιδίους πόρους και σας το λέω αυτό διότι εάν ναι, συμβάλλει ο χρηματοοικονομικός ε, τομέας, αν βασιστούμε στη δική του ε, συμβολή, θα πρέπει ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε και έναν έλεγχο ε, αυτού του Κορβανά επίσης ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το κονδύλι είναι επαρκές αλλά όχι υπερβάλλον. Ε, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν ίδιους πόρους ε, οι εποπτικές αρχές για λόγους ανεξαρτησίας και ο κύριος Σάντσες Πρεσέντο έχει απολύτως δίκιο στην εκθεσή του και θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Ευχαριστούμε λέει ο κυρία Γένσεν, ο δόκτωρ Χάνς Πίτερ Μάρτιν τώρα. Um, Ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι παλιό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και έχω μερικές παρατηρήσεις που έχουν να κάνουν με την ε, απαλλαγή των διαφόρων οργανισμών. Ε, ο κύριος Λάγκεν πέρσι ήταν συγητής και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει, υπήρχε πρόβλημα στο κόστος από τη λειτουργία και τη δομή. Ήταν τεράστια τα μισθώματα ας πούμε που έπρεπε να καταβάλουν. Και με τα μισά λεφτά κανονικά θα μπορούσαν να είχαν βρει αντίστοιχα γραφεία. Ε, ρωτώ λοιπόν, τι απέγινε, ε, βγήκαν τίποτα συμπεράσματα, υπήρξαν συνέπειες από αυτές τις περσινές παρατηρήσεις. Και ένα δεύτερο, που έχει και αυτό να κάνει με οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεσμικά όργανα για την απαλλαγή. Συστηματικά ε, ρωτούσαμε τι γίνεται με το κόστος μετάφρασης για την εσωτερική μετάφραση που γίνεται από υπαλλήλους. Και επικεφαλής εκεί είναι το ελεγκτικό συνέδριο για λόγους μυστήριους σε μας. Όλα τα μεταφράζουν προς τα γαλλικά στο Λουξεμβούργο, στο ελεγκτικό συνέδριο. Μέχρι 341 ευρώ, επαναλαμβάνω, 341 ευρώ κοστίζει σελίδα. Και ζήτησα να συγκριθεί με τις τιμές της αγοράς και διεθνώς, που είναι πολύ υψηλού επίπεδου και βεβαίως υπάρχουν και έγγραφα πάρα πολύ απόρριτα, αλλά όλα αυτά κινούνται γύρω στα 100 ευρώ. Και αυτό είναι πραγματικά μια στρεβλή κατάσταση που ισχύει και σε άλλα θεσμικά όργανα. Και ρωτώ τον εισηγητή και για τις νομοδοτήσεις προβλέπετε τίποτα για στα πλαίσια των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για τα οποία εμείς νομοδοτούμε να υποδείξουμε αυτό το θέμα γιατί είναι συνολικά εκατομμύρια ευρώ ή μήπως δεν είναι κανένα θέμα αυτό για μας και δεν μας απασχολεί. Ευχαριστώ. Η κυρία Λούλη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Ήθελα μόνο να πω ότι έχω κάποιους ενδιασμούς ε, για το, αυτό που αναγράφεται στο σημείο 2. Ε, όταν μιλάμε ε, για την ΟΝΕ ε, ναι και για τη μελλοντική χρηματοδότηση θα έλεγα ότι ε, καλό θα ήταν να πούμε ότι χάρη στις αρχές συμβάλλουμε στη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών που είναι απαραίτητη για την οικονομική μεγέθυνση και ως εκ τούτου της ε, δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας όμως δεν είναι αυτός καθ' αυτός ο ρόλος τους να οργανώσουν δηλαδή την ανάκαμψη της οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Θα πρέπει λοιπόν να ε, τροποποιήσουμε λίγο τη χρειά τη φαρασιολογίας που χρησιμοποιούμε για τον προπολογισμό. Ε, ναι, θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ε, Θα συμφωνήσω παρόλα αυτά ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, πρέπει να χρηματοδοτηθούν οι υποπτικές αρχές στα πλαίσια του προϋπολογισμού της Ένωσης και όχι στα πλαίσια του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάποιος ε, αναφέρθηκε στην έκθεση Giggold Εγώ είμαι σκιώδης εισηγήτρια, δεν είδα όμως παρόλα αυτά μέχρι στιγμής συμβαστικέ προτάσεις από πλευράς του κυρίου Γκίγκολτ. Εγώ το μόνο που ζητώ είναι στην Επιτροπή μας να μην λέμε κάτι στην έκθεση Γκίγκολτ και το αντίθετό του στην έκθεση Πρεσέντο. Νομίζω ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε κάποια συνέπεια. Ήδη οι είναι ένα άλλο ζήτημα που αναφέρθηκε, δηλαδή η χρηματοδότηση από τις τράπεζες και από τους εποπτευόμενους. Ε, εδώ θα πρέπει να αποφύγουμε ε, την ε, επικάλυψη. Ήδη σε εθνικό επίπεδο οι τράπεζες, οι εποπτευόμενοι, Ε, ήδη ε, χρηματοδοτούν. Τουλάχιστον ε, αυτό συμβαίνει στο Λουξεμβούργο. Δεν θα πρέπει λοιπόν να επιδιώξουμε διπλή χρηματοδότηση, κυρίως σεβόμενοι και τους κανόνες λειτουργίας της ΟΝΕ. και όντως θα πρέπει να ελέγξουμε τα έξοδα προσωπικού και να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν ε, τα απαιτούμενα κονδύλια. Αλλά δεν συμφωνώ να πούμε απλώς ότι πρέπει να αυξήθουν, να πούμε ότι τα κονδύλια για τον προπολογισμό γενικότερα και ειδικότερα για το προσωπικό θα πρέπει να αυξηθούν ε, όπου δει, όχι γενικότερα. Θα καταθέσω και σχετικές ε, τροπολογίες. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις που ήθελα να κάνω. Ευχαριστώ κυρία Λούλινγκ. Αν δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο, θα δώσω το λόγο ξανά στον εισηγητή, τον κύριο Σάντς Πεσέδα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλες τις παρεμβάσεις και υποδείξεις. Παρακολούθησα την, ε, τον όλο διάλογο και θα ήθελα να σχολιάσω ε, ορισμένα ζητήματα ως προς τους ε, ορισμούς. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών ε, αφορούν το τραπεζικό σύστημα και θα πρέπει να είναι φερέγγοι οι οργανισμοί, δηλαδή να εγγυώνται μάλλον την φερεγγιότητα. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη την ε, ανάκαμψη της αγοράς μέσα στα πλαίσια μιας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση του, του ζητήματος της κρίσης. Για να φτάσουμε αυτούς τους στόχους θα πρέπει να πληρούν το, το ρόλο τους και τα καθήκοντά τους. Σε σχέση με τους ε, ορισμούς μέσα στα πλαίσια του καθεστώτος εποπτείας και των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το στάδιο αυτό των εργασιών και διεργασιών. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο σχεδιασμός και διαχείριση των χρηματοοικονομικών μέσων με επάρκεια, με διαφάνεια και γι' αυτό όλες οι τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση είναι ευπρόσδεκτες. Θα ήθελα να πω ότι ότι ε, περιορίστηκα στο 2012 στην απαλλαγή για αυτό το οικονομικό έτος. Ε, ίσως για άλλα υπάρχουν άλλες διαδικασίες με βάση την εισήγηση το, του ελεγκτικού ε, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η διαφάνεια για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή το ελεγκτικό συνέδριο στην έκθεσή του έφυξε και άλλα ζητήματα τα οποία όμως δεν συμπεριέλαβα. Αν πρόκειται όμως για το ε, ημερολογιακό έτος 2012 θα συμπεριλάβω όλα όσα χρειάζονται. Μέσα στα πλαίσια των χρηματοοικονομικών μέσων και πόρων που διατίθενται θα πρέπει να δούμε τι βελτιώσεις μπορούν να επέλθουν και όλο το σύστημα, το όλο σύστημα των πόρων θα πρέπει να είναι ένα συνεκτικό ζήτημα με βάση ε, τη λειτουργία αυτών των αρχών. Κάτι το οποίο προωθεί η Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις σας. Ελπίζω να λάβω και τροπολογίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις πτυχές που μας απασχολούν στην Επιτροπή μας. Ευχαριστούμε πολύ Αντολή. Προθεσμία, η προθεσμία λήγει στις 22 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι υποβολής τροπολογιών και στις 3 ε, Φεβρουαρίου, 13 Φεβρουαρίου θα συζητηθεί ε, η έκθεση και η τελική ψηφοφορία θα γίνει στις 18 Μαρτίου. Περνάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι το 7. Σύμφωνη συνεργασίες Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή της πολιτικής του ανταγωνισμού. Ο εισηγητής είναι ο κύριος Κούτας, ο οποίος έχει και το λόγο. Thank you, thank you, Pablo. Since it's the first time, let me wish you all of you happy. Σας εύχομαι καλή χρονιά. Καταρχήν και τώρα σε σχέση με το θέμα μας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις τροπολογίες που έχουν υποβάλει. Νομίζω ότι βελτιώνουν το κείμενο. Χτες είχαμε μία συνάντηση των σκιωδών. Δεν ανέκυψαν σημαντικά ζητήματα ως προς τις τροπολογίες. Νομίζω ότι θα επιτευχθεί μεγάλη πλειοψηφία. πιο σημαντικό ζήτημα είναι το χρονοδιάγραμμά μας, γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας γενικότερα και θα πρέπει να επέλθει αυτή η συμφωνία. Είναι προς ε, ίδιο συμφέρον. Για την 1η Φεβρουαρίου, μάλλον ο προγραμματισμός προβλέπει την 1η Φεβρουαρίου ως ε, καταληκτική ημερομηνία. I Δηλαδή, κατά τη γνώμη πρέπει να συζητήθει στην πρώτη σύνοδο του Φεβρουαρίου στην Ολομέλεια. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε και το χρονοδιάγραμμα ε, όπως προβλέπεται μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας μας ε, με την Ελβετία και θα ήθελα να συμφωνήσουμε στην ΕΚΟΝ καταρχήν και θα δούμε Ε, πώς θα διαμορφωθεί και η πρόταση ψηφίσματος με βάση την έκθεση. Θα ήθελα να μάθω τις, να, να μου μάλλον υποβάλλετε προτάσεις και υποδείξεις σε σχέση με την αρχική αυτή πρόταση και για τις τροπολογίες και θα δεχτώ να γίνουν μικρές, μικρές ε, διευθετήσεις και προσαρμογές αν είναι αναγκαίο. Ευχαριστούμε κυρία Κούτα, έξω ονόματος του, ε, του ΕΛΚ, ε, ο κύριος... Merci. Σε αντικαθιστά τον κύριο Μάρκους Φέρμπερ. Ευχαριστώ. Ο Μάρκους Φέρμπερ. Ο κύριος Γκοζές, με συγχωρείτε. Ο κύριος Μάρκους Φέρμπερ μου υπέβαλε ε, ένα κείμενο και το οποίο θα σας αναπτύξω. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει ε, κάποια μεγάλη διαφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων και θα φτάσουμε σε μία καλή ποιοτική συμφωνία. Υποστηρίζουμε την συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελβετίας, διότι έτσι θα βελτιώσουμε τις δυνατότητες συνεργασίας μέσα στα πλαίσια της πολιτικής ανταγωνισμού μεταξύ αρμοδίων αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελβετίας. Εξάλλου αυτή η συμφωνία συνεργασίας ανοίγει το δρόμο για άλλες συμφωνίες και το ΕΛΚ υποστηρίζει την πρόταση αυτή Άρα θα υποστηρίξουμε τις τροπολογίες συμβασμού που θα προτείνει ο εισηγητής, όμως υπάρχουν δύο τροπολογίες που δεν θα δεχτούμε, που αφορούν την φορολογική εναρμόνιση, που δεν θεωρούμε ότι αφορά ε, ζητήματα που άπτονται της έκθεσης αυτής. Ως προς το χρονοδιάγραμμα θα θέλαμε να ακολουθήσουμε μια τάχη στη διευθέτηση εν ευθέτω χρόνο και εάν μέσα στα πλαίσια ε, της ε, παράλληλης γνωμοδότησης η Ελβετία ε, δεν αντιτάξει κάτι σημαντικό θα μπορέσουμε να δεχτούμε και μία προφορική τροπολογία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Θα θέλαμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα και τους στόχους που έχουν οριστεί. Ευχαριστώ, πολύ κύριε Γκοζές. Εξ ονόματος τώρα των φιλελευθέρων, ουδής, διότι απουσιάζω. Φαντάζομαι δεν θα θέλει κανείς φιλελεύθερος να μιλήσει. Ε, ο κύριος Λάμπερτς ε, είναι ε, κανονικά ο σκιώδης των Πρασίνων, αλλά έχει αντικαταστάτη. είναι ο κύριος Μπεσέ. ο, συνάδελφος και φίλος Φιλίπ Λαμπέρτς δυστυχώς κολλείεται και ζητεί συγγνώμη για την απουσία του. Τον αντικαθιστώ εγώ. Να πω με δύο λόγια τα εξής. Η ομάδα μας υποστηρίζει ε, τη γραμμή του εισηγητού, ε, τις συμβαστικέ προτάσεις που μας διαβιβάστηκαν πρόσφατα, καθώς επίσης και τις περισσότερες τροπολογίες που ε, κατετέθησαν από τους κοιότητες εισηγητές. Παρόλα αυτά, έχουμε μια μικρή επιφύλαξη πολιτική ως προς τις προτεραιότητες, πάντα τις πολιτικές προτεραιότητες. Λυπούμεθα που τα θέματα του αθέμη του ανταγωνισμού ε, κυρίως στη φορολογία και μάλιστα ο εταιρικός φόρος δεν ε, εξετάζεται εδώ. Γίνονται έρευνες αυτόν τον καιρό από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού ως προς ε, ορισμένα φορολογικά συστήματα στην Ιρλανδία, κάτω χώρες και στο Λουξεμβούργο και δείχνει ότι υπάρχουν σαφέστατα προβλήματα σε σχέση με αυτά παρόλο που γνωρίζουμε ότι ο θέμητος ανταγωνισμός δεν σταματά στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, λυπούμεθα γενικότερα, θα επιθυμούσαμε να ε, αναφέρεται και στη διάσταση αυτή η έκθεση. Αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υποστηρίζουμε την πρόταση του εισηγητού ίσα ίσα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βεσέ, εξ ονόματος ε, των συντηρητικών ουδής, εξ ονόματος των ε, της ΓΟΕ, κύριος Κλούτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν επιθυμεί να μιλήσει, θα της δώσουμε το λόγο. Pues nada, entonces, ε, Λοιπόν, καλά. Όχι, πρέπει να ξαναμιλήσει ο εισηγητής. Συγγνώμη, είμαι λίγο φερημένο σήμερα. Thank Παύλο, θέλω να απαντήσω μόνο στον ε, κύριο Μπεσέ. Ναι, να υποστηρίξω αυτές τις τροπολογίες ε, για τη φορολογία, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι στο σωστό σημείο, στο σωστό φάκελο. Εδώ συζητούμε για ανταγωνιστικότητα. Είμαστε, είναι λίγο εκτός θέματος. Σε κάθε περίπτωση δεν είμαι κατά ανθρωπολογιών του κύριου Λάμπερτς. Ευχαριστώ κύριε Κούτας. Κύριε Λούλινγκ. Euh, κύριε Πρόεδρε, ήθελα μόνο να πω πως πρέπει να ε, σταματήσουμε επιτέλους να επιτιθέμεθα ε, στα κράτη-μέλη για το φορολογικό του σύστημα. Ε, είναι θέμα επικουρικότητας. Εκτός μικρόφωνου το σχόλιο. Ε, όχι, ε, βαρέθηκα πια. Να έρθουν στο Λουξεμβούργο για να δουν αν είναι φορολογικός παράδεισος. Δεν ισχύει αυτό. Εμείς ανέκαθεν ήμασταν υπέρ του ε, θεμητού ανταγωνισμού ακόμη και φορολογικά ζητήματα. Και όλα είναι αλληλένδετα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το θέμα μας το βασικό δεν είναι τα φορολογικά. Μιλάμε για την πολιτική ανταγωνισμό. Και αυτό δεν υπάρχει στη δική μας αρμοδιότητα. Ε, άμα ήταν ε, έκθεση της Επιτροπής Γυναικών ε, θα μιλούσαμε και για την άμβλωση μέσα στην έκθεση ανταγωνιστικότητας. Όλα τα είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μείνουμε εντός θέματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λούλινγκ για τα σχόλια αυτά και προχωρούμε. Στις 20 Ιανουαρίου θα ψηφίσουμε την έκθεση αυτή στην Επιτροπή μας, ενώ στην Ολομέλεια, στη δεύτερη Σύνοδο Ολομελίας του μηνός Φεβρουαρίου. Επόμενο θέμα στη Μεσαία Διάταξη. Υπαριθμόν 8. Ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια. Έχει αναβληθεί η συζήτηση για το θέμα αυτό και τώρα κανονικά και θεωρητικά θα έπρεπε να περάσουμε στο σημείο 9 που ε, αφορά την ε, εξέταση των τροπολογιών της εκθέσεως ε, για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας με εισηγητή τον κύριο Βολφ Κλίντς, ο οποίος είναι καθοδόν μου λέει η γραμματεία, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα μέχρι να έρθει ο κύριος Κλίντς. Ε, Επαναλαμβάνεται η διακοπή σας συνεδρίαση. Σημείο 9. Μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Εξέταση των τροπολογιών. Η συγητής είναι ο κύριος Κλίντς, ο οποίος και κατέφθασε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφε που μου δίνετε το λόγο. Βλέπω ότι Αποσιάζουν και ορισμένοι σκιώδεις ηγητές. Φαίνεται ότι τα ξεπετάξατε σήμερα τα θέματα πρωί-πρωί, γιατί είχε προβλεφθεί για αργότερα το θέμα. Οι τροπολογίες που κατατέθησαν είναι 150 και πλέον συνολικά. Ε, πρέπει να σας πω ότι διαβάζοντας και μελετώντας τις τροπολογίες διαπίστωσα ότι υπάρχουν πολλές ε, ε, που συμφωνούν με την ουσία των πραγμάτων και την οπτική γωνία. Μπαίνω λοιπόν στη συζήτηση αισιόδοξο, ε, ε, συζήτηση όχι μόνο με τους κοιόδης αλλά και με άλλους συναδέλφους και πιστεύω ότι την άλλη εβδομάδα ήδη θα μπορέσουμε να έχουμε συμβιβαστικές προτάσεις για να υποβάλουμε στους σκιώδες ηγητές και να αποτελέσουν ε, αυτές τη βάση για μια συμφωνία. Οι πάντες συμφωνούν ότι η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι ουσιαστικό στοιχείο και της οικονομικής πολιτικής της Ένωσης και των κρατών μελών και θα συνεχιστεί αυτό και στο μέλλον. Η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση σημαντικών ε, προγραμμάτων και έργων, ιδιαίτερα υποδομών, ενέργειας, ανάπτυξης, που ε, αποτελούν βασικά βασικές προϋποθέσεις για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διατηρηθεί αυτή και για να βελτιωθεί όπου αυτό είναι δυνατό. Το θέμα λοιπόν αυτό κυριαρχεί ή κανονικά θα πρέπει να κυριαρχεί ε, στην προοπτική των επομένων ετών και στον προβληματισμό. Στην Ευρώπη έχουμε συνηθίσει η χρηματοδότηση ε, παντός είδους και οι μακροπρόθεσμη ε, οι επενδύσεις να έρχονται από τις τράπεζες. Σε αντίθεση με τις Ηνωμένε Πολιτείες που η συμμετοχή της τραπεζικής χρηματοδότησης είναι χαμηλότερη, εμείς είμαστε στο 75%. Με την κρίση λοιπόν και την παγκόσμια οικονομική κρίση και τις επόμενες ε, και προκλήσεις για τις τράπεζες αλλά και με τα αριθμιστικά μέτρα οι ε, χορηγήσεις των τραπεζών και οι δανειοδοτήσεις έχουν δυσκολευτεί. Δηλαδή χρειάζεται υποστήριξη από ίδια κεφάλαια περισσότερα. Υπάρχει και κατάσταση του χρέους στα περισσότερα κράτη-μέλη, οπότε η κλασική μορφή χρηματοδότησης δια του τραπεζικού τομέα στο μέλλον δεν παρκεί πλέον. Θα πρέπει να αναζητήσουμε νέους δρόμους και να βρούμε κυρίως νέους δρόμους και τρόπους για να εξασφαλίσουμε τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Μόνο με μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση καλών και ουσιαστικών προγραμμάτων θα καταφέρουμε να ξαναφέρουμε την Ευρώπη σε λογικούς ρυθμούς ανάπτυξης και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας τις οποίες θα εξασφαλίσουμε κιόλας. Τι διαπιστώνουμε. Στην Ευρώπη γενικότερα και συνολικά είναι χαμηλή η προθυμία ανάληψης κινδύνου. Δεν ρισκάρουμε. Οπότε όλη αυτή η χρηματοδότηση που ενέχει ένα κίνδυνο δεν κυριαρχεί όπως σε άλλες περιοχές του κόσμου, όπως στη Βόρεια Αμερική κυρίως, και θα πρέπει να καταφέρουμε τα επόμενα χρόνια να κάνουμε κάτι παραπάνω για να ε, τονώσουμε αυτή την κουλτούρα και αυτή την προθυμία ε, να αναλαμβάνει κανείς κίνδυνο στη χρηματοδότηση. Να υπάρχει μια τολμηρή, ας πούμε, ε, νοοτροπία. Έχουν γίνει τροπολογίες και να μπω σε αυτές και στις προτάσεις των συναδέλφων. Σχεδόν όλοι όσοι υπέβαλαν τροπολογίες αναφέρονται στο θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και φαίνεται ότι όλοι έχουν προβληματιστεί για το πώς θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, με τρόπο πιο εύκολο και λιγότερο γραφειοκρατικό. Να έχουν ε, στη διάθεσή τους τα κονδύλια που χρειάζονται για να υλοποιούν τα επιχειρηματικά τους σχέδια και να αναπτυχθούν να αξιοποιούν τις ευκαιρίες ανάπτυξης που τους ανοίγονται. Είναι καλές οι προτάσεις αυτές των συναδέλφων και θα ε, καταβάλουμε προσπάθειες ε, στις συμβασικές τροπολογίες να αναφερθούμε αναλόγως και στις μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις. Ένα άλλο θέμα είναι κάτι που στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει ε, ε, υποστεί ε, πολύ αρνητική εικόνα. Αφορά αυτό την τιτλοποίηση. Ας πούμε, με την κρίση των subprimes στις Ηνωμένε Πολιτείες έχει λάβει μία αρνητική χρειά αυτό αλλά δεν θα πρέπει μαζί με τα, χλωρά, με τα ξερά να καίγονται και τα χλωρά. Έχει γίνει με ένα στρεβλό τρόπο αυτή η τιτλοποίηση. Ε, τα στοιχεία του ενεργητικού ε, ε, πολύ συχνά είχαν υποστηριχθεί από λανθασμένες εκτιμήσεις των οίκων αξιολόγησης, αλλά δεν είναι κάτι που πρέπει να εγκαταλειφθεί τελείως αυτό. Απλώς θα πρέπει να γίνεται με το σωστό τρόπο το έχει αποφασίσει και το Κοινοβούλιο, δηλαδή με άλλα λόγια να υπάρχει ένα ε, ε, στοιχείο ε, διακράτησης ίδιο και να μην υπάρχουν πάρα πολλά κλιμάκια. Δηλαδή να μην έχουμε τιτλοποίηση, επιτιτλοποίησης να σπάνε συνεχώς τα προϊόντα σε μικρότερα μερίδια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται από τους συναδέλφους και έχουν δίκιο να εκπονήσει έναν ορισμό για το τι εστί, τιτλοποίηση υψηλής ποιότητας, ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει και ποια μορφή. Και εμείς ε, πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική ε, Τράπεζα ε, με το International Financial Stability Board να ασχοληθούν με αυτό τον ορισμό. Ένα τελευταίο που θέλω να αναφέρω λοιπόν είναι οι φόροι. Οι φόροι ξέρουμε ότι είναι ε, εξουσία και αρμοδιότητα των κρατών μελών και το γνωρίζουμε και ξέρουμε ότι δεν πρόκειται πολύ γρήγορα να το αλλάξουμε. Αφήστε δε που δεν είναι απόλυτη η πρόθεσή μας πάντα. Αλλά το φορολογικό πλαίσιο παίζει ρόλο, ιδιαίτερα και πάλι στην προθυμία θεσμικών επενδυτών αλλά και ε, ιδιωτών επενδυτών να ε, επενδύουν μακροπρόθεσμα. Έχω υπόψη μου ένα παράδειγμα από την Allianz που είναι μεγάλη γερμανική ασφαλιστική εταιρεία και η οποία αποφάσισε στη Νορβηγία να επενδύσει σε ένα μεγάλο έργο υποδομής. Όπερ και Εγένετο. Ε, και υποθέτοντας θεωρώντας ότι θα υπάρχει μια συγκεκριμένη φορολογική μεταχείριση για αυτό το έργο. Έκανα την επένδυση αυτή και δύο χρόνια μετά ανετράπη εκβάθρων αυτό το φορολογικό πλαίσιο και η βάση για την καταρχήν θετική απόφαση ε, κατακριμνίστηκε. Δηλαδή, αν είχε αλλάξει το φορολογικό σύστημα και το ήξερε η εταιρεία πριν από δύο χρόνια, δεν επρόκειτο ποτέ να είχε κάνει αυτή την επένδυση στην Νορβηγία. Προσοχή λοιπόν χρειάζεται εδώ. Χρειαζόμαστε αξιόπιστα φορολογικά συστήματα, φορολογικά πλαίσια με διαφάνεια που να ισχύουν για ένα μακρύ χρονικό διάστημα και μπορεί κανείς να είναι πεπισμένος και να υπαφίδει σε αυτό. Γιατί εδώ πρόκειται για μακροπρόθεσμες επενδύσεις, οπότε είναι πάρα πολύ αποφασιστικό να μην ανατρέπονται τα δεδομένα στη μέση της επένδυσης και μάλιστα πολύ νωρί μετά την επένδυση. Επίσης κάτι άλλο πολύ σημαντικό, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει διπλή φορολόγηση σε δύο χώρες και περισσότερες. Και επίσης δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να υπάρχει διπλή φόρο αποφυγή ή αφορολόγητο. Μας μας ενδιαφέρει τα κράτη-μέλη να εισπράττουν τους φόρους που δικαιούνται και τους αναλογούν και να μην υπάρχουν ε, διάφορα τεχνάσματα ή ε, δυνατότητες και παραθυράκια ώστε να μην πληρώνει πουθενά σε καμιά χώρα ε, ο επενδυτής επικαλούμενος τη μη διπλή φορολόγηση. Αυτά και περιμένω τα προφορικά σχόλια των συναδέλφων Έχουμε ήδη συμφωνήσει να βρεθούμε στο Στρασβούργο με τους και ηγητές σε μια συνεδρίαση και ελπίζω τελικά να προχωρήσουμε με καλό τρόπο και ουσιαστικό και να βάλουμε τα θεμέλια για την τελική εκδοχή της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ. του Ο κύριος Γκοζές έχει το λόγο εξ ονόματος του κυρίου Αλφρέντο Παλών. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είμαι ένα σε τρεις. Τρεις σε έναν μάλλον. Τώρα έχω το καπέλο του φίλου Αλφρέντο Παλώνε. Ε, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί δυστυχώς και θα ήθελε να σας διαβιβάσω δύο μηνύματα. Καταρχήν ε, να ευχαριστήσει τον εισηγητή και το κάνω και εγώ γιατί πρόκειται για τον Βόλφ. Και δεύτερον μία συμφωνία γενικά στη, με τις τροπολογίες δεν έχει κάποιο μείζον ζήτημα. Θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση των σκιωδών που προβλέπεται στην ημερομηνία που είπε ο Βόλφ. Ευχαριστούμε κύριε Γκοζές εξ ονόματος των σοσιαλιστών. Ε, ο κύριος Κούτας ε, έχει το λόγο, αντικαθιστώντας κάποιον άλλον, τον κύριο Λιέμ Χονγκ Νιόκ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή για, την, ε, για το σχέδιο έκθεσης που αποτελεί μια πολύ καλή βάση ε, εργασίας. Έχει υποβάλει μια σειρά τροπολογιών έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη καλύτερα η ένα του μακροχρόνιου επενδυτή και δημόσιου μακροχρόνιου επενδυτή ιδιαίτερα. Έτσι ώστε να υπάρχει μία ε, προβλεψιμότητα φορολογική και δικαιοδοτική. Οι δημόσιοι μακροχρόνιοι επενδυτές όπως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ε, τοπικά, περιφερειακά και μη, θα διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο μακροχρόνια και γι' αυτό θα πρέπει τα κράτη-μέλη να προωθήσουν αυτή τη συνεργασία όπως ορίζει την τροπολογία 73 και ως προς τις ΜΜΕ θα πρέπει να προβλέψουμε ε, ορισμένα βασικά στοιχεία, δηλαδή να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην αγορά ε, κεφαλαίου και η τροπολογία 99 αυτό ακριβώς ορίζει ότι η ΕΤΕ θα πρέπει να προβλέψει συγκεκριμένα μέτρα για τις ΜΜΕ. Επίσης, θα πρέπει να ε, υπάρχει σωστή χρήση τιτλοποιημένων προϊόντων. online. θέλει να τονίσει ότι η τιτλοποίηση είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες αντιμετώπισης της χρήσης και θα πρέπει να χειριστούμε ανάλογα. Η έκθεση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ε, για να επιτρέψει την μαζική τιτλοποίηση στην ε, ε, αγορά και στην τροπολογία 19 τονίζει ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε ε, μία σωστή διατύπωση έτσι ώστε να ε, έχουμε μία σωστή ρύθμιση στη διαδικασία τιτλοποίησης. Ο Λάιμ πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρχει η ύψιστη δυνατή διαφάνεια και η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού ε, Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας. Ο ΛΑΙΜ επίσης στην 131 επί της παραγράφου 26 προωθεί ε, συγκεκριμένα μέσα για τους θεσμικούς επενδυτές έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα ε, πρότυπα για να μην υπάρχει πτυτικότητα της αγοράς, να μειωθεί δηλαδή ο ΛΑΙΜ πιστεύει ότι θα φτάσουμε σε πολύ καλές προτάσεις συμβιβασμού και θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την πράσινη βίβλο της Επιτροπής μέσα στα πλαίσια του καθεστώτος ρύθμισης μακροχρόνιων επενδύσεων. Στην Ευρώπη ευχαριστούμε. Εξ ονόματος των Πρασίν, ο κύριος Μπεσέτ έχει το λόγο. Ε, αντικαθιστώντας τον κύριο Άικαουτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο συνάδελφος ε, δυστυχώς ε, είναι στην Ολλανδία, δεν μπόρεσε να προσέλθει και θα ε, ήθελε να σας πω ότι στη συνάντηση σκιωδών του Στρασβούργου θα παρευρεθεί. Τώρα, ως προς ε, τις δικές μας τροπολογίες, θέλουμε να εμπλουτίσουμε την εξαιρετική έκθεση του κυρίου Κλίντς, εμείς Θέλουμε να κινηθούμε προς ε, τρεις κατευθύνσεις. Καταρχήν ε, να ενσωματώσουμε το περιβάλλον, την ενέργεια και το κλίμα σε αυτή την έκθεση μέσα στα πλαίσια των μακροχρόνιων επενδύσεων. Και αυτός είναι και ο στόχος των τροπολογιών μας. 49 και 129 ιδιαίτερα. Θα πρέπει να λάβουμε ε, υπόψη τους ε, βραχυπρόθεσμους και μακροχρόνιους ε, κινδύνους, ακριβώς επειδή υπάρχει μεγάλη συσσόρευση άνθρακα, κάτι το οποίο ε, δεν μας ε, οδηγεί στο να αντιμετωπίσουμε τους ε, κλιματικού μας, κλιματικούς μας στόχους. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει κατάλληλη ρύθμιση για να διευκολύνουμε τις μακροχρόνιες επενδύσεις που θα οδηγήσουν σε εξωτερικές αναθέσεις, δηλαδή σε ευρωπαϊκές δέκο. Η ομάδα μας θέλει να ενθαρρύνει μία οικονομική μακροχρόνια αξιολόγηση έτσι ώστε να εντάξουμε αυτούς τους παράγοντες σε σαφείς παραμέτρους λαμβάνοντας υπόψη τα μακροχρόνια ε, επενδυτικά σχέδια των δημοσίων αρχών και μέσα στα πλαίσια των ομολογιών έργων. Η τρίτη πτυχή, τονίζει ο Σκιώδης, έχει ως εξής θα θέλαμε να ε, λάβετε υπόψη την τροπολογία 93 που υπέβαλε, που θεωρεί ότι είναι ένας πολύ καλός συμβιβασμός με βάση τις θέσεις που έχουν ε, εκτεθεί ως προς την τιτλοποίηση μέσα στα πλαίσια των ε, μακροχρόνιων πεντήσεων καθώς και την 87 που τονίζει τους καινοτόμους μηχανισμούς ιδιαίτερα το, τη χρηματοδότηση και τη δανειοδότηση μεταξύ ομοτήμων. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπεσέτ. Ο κύριος Καμάλ θα λάβει το λόγο εξ των Ευρωπαίων Μεταρρυθμιστών και Συντηρητικών. Φαίνεται ότι μόνο ο κύριος Κλίντς μιλάει εξ ονόματός του. Όλοι οι άλλοι έχουν αναθέτουν σε κάποιον άλλον. Εγώ εκπροσωπώ τη Βίκη Φόρτ σήμερα λοιπόν ε, ίσως σας απογοητεύσει αυτό και όποιος γνωρίζει τη Βίκη ξέρει ε, ότι, ε, ότι πάντα ε, προβάλλει συγκεκριμένες θέσεις αναλυτικά. Εγώ θα το κάνω συνεκτικά. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κλίνς και συμμερίζεται τις ανησυχίες σε σχέση με τις, με τις μακροχρόνιες επενδύσεις και τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις. Θα πρέπει να αρθούν ορισμένα ε, στοιχεία της νομοθεσίας, το οποίο, τα οποία έχουν ολέθριες συνέπειες, ιδιαίτερα σε σχέση με το φορολογικό καθεστώς, διότι ε, οι φόροι σημαίνουν ότι πολλές φορές έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα ή αντίθετα όχι. Ας πούμε το FTT κινείται προς αυτή την κατεύθυνση γιατί ξέρουμε ότι το εμπλεκόμενο κόστος περνάει στους επενδυτές. Βεβαίως υπάρχει και το θέμα της ε, διπλής ε, φορολόγησης, όπως είπε και ο κύριος Κλίνς. Δεν θεωρεί ότι η νέα νομοθεσία είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των ε, μακροχρόνιων επενδύσεων. Φόρτ ασχολήθηκε με ιδιαίτερες τροπολογίες που αφορούν τη δημόσια, τις δημόσιες επενδύσεις. Θα πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη πώς χρησιμοποιούνται τα χρήματα του φορολογούμενου Βεβαίως, ε, στον τομέα των υποδομών ε, της ενέργειας και υγείας θα πρέπει να επενδύσουν οι δημόσιοι επενδυτές, αλλά το κράτος δεν διαθέτει τα χρήματα πολλές φορές. Γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους ιδιωτικούς επενδυτές και να ε, γίνει αυτό στο σωστό ε, περιβάλλον. Επίσης θα πρέπει να προωθήσουμε εταιρικές σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η κυρία Φόρτ καλωσορίζει τις τροπολογίες ε, βελτίωσης της θέσης των ΜΜΕ και θεωρούμε ότι υπάρχει συνένεση και εδώ και σε αυτή την Επιτροπή και σε άλλες υπέρ των ΜΜΕ η παράγραφος 25 θα πρέπει να διαγραφεί σε σχέση με τις επενδύσεις ε, υποδομών. Θεωρεί ότι δεν είναι σκόπιμο και θεωρούμε ότι θα πρέπει το θέμα αυτό να προωθηθεί σε τριμερείς διαλόγους και όχι εδώ. Άρα θα πρέπει να ε, διαγραφεί η παράγραφος 25. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για την οδηγία κεφαλαιακών απαιτήσεων ή επάρκειας. Όπως καταλαβαίνετε, η ομάδα μας δεν είναι υπέρ της φορολογικής εναρμόνισης και δεν θεωρούμε ότι θα έδινε κίνητρα για μακροχρόνιες επενδύσεις. Θα, ε, θέλαμε να κάνουμε μία έκκληση και προς τον κύριο Κλίντς να συμπεριλάβει ορισμένες τροπολογίες της Vicky Ford. Δηλαδή ε, ως προς την ε, διαδικασία πτώχευσης θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ε, μια καλύτερη θεώρηση αλλά θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει ομογενοποίηση του καθεστώτος. Επίσης θεωρούμε ότι θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα το ζήτημα μέσα στα πλαίσια της γενικότερης χρηματοδότησης με τη συνέργεια ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Ως προς την τιτλοποίηση, η δίκη θα ήθελε να υπάρξει ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας της ε, τιτλοποίησης. Θεωρούμε ότι ε, πρόκειται για έναν άλλον χρηματοοικονομικό εφημισμό. Δηλαδή, ε, μιλάμε για πράξεις υπέρ των περιουσιακών και κινητών στοιχείων που δεν βοηθούν παρά τις, ε, τους οργανισμούς πιστοληπτικής ικανότητας έτσι ώστε να χορηγήσουν ένα τριπλό α και τίποτα άλλο. Και αυτά είναι ένα από τα διδάγματα της κρίσης από τα οποία θα πρέπει να αντιλήσουμε κάτι το συγκεκριμένο, δηλαδή πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της τιτλοποίησης. γιατί πολλοί χρειάστηκε να ασχοληθούν με τα CDS για έξι μήνες πριν καταλάβουν ποιο είναι το λανθάνον χρέος που βρίσκεται πίσω από αυτό. Εάν γίνει καλή χρήση της τιτλοποίησης, τότε θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το, τις μακροχρόνιες επενδύσεις. Θα θέλαμε να σας ευχαριστούμε και η Βίκη και εγώ. Ευχαριστούμε κυρία Καμάλ. Από τους πράσινους, ο κύριος Χάντελ, ο οποίος δεν είναι παρόν. Α, με συγχωρείτε, της Γκουε, της Γκουε. Ο κύριος Χάντελ δεν ξέρω κατά πόσο κάποιος μπορεί να τον αντικαταστήσει. Φαίνεται πως όχι. Η κυρία Λούλινγκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συγητή, τον Βολφ Κλίντς. Είμαι η μοναδική πλέον, εκτός από τον ίδιο, που μιλώ εξ ονόματός μου εδώ. Που είμαι η ίδια παρούσα. Αυτό έχει να κάνει με τις πέμπτες γενικά. Ε, ε, ε, οι Λουξεμβούργοι με τα γερμανικά, γαλλογερμανικά που μιλάνε το λένε αψαντεΐσμους που είναι η κοπάνα ουσιαστικά. Τα μισά γαλλικά, τα μισά γερμανικά. Είναι πολύ σημαντικές επιτροπές και θα πρέπει να ορίζονται εδώ μέλη που να ξέρουν ότι η δουλειά τους είναι εδώ, στις Βρυξέλλες. Και τις πέμπτες ξέρετε οι υπόλοιποι πολίτες έχουν εβδομάδα πέντε ημερών, Εμεί την κάναμε τεσσάρων ημερών, ε, γιατί τέσσερι ημέρες συνεδριάζουμε, αλλά πέντε μέρε μπορούμε και να δουλεύουμε, δεν πειράζει. Λυπάμαι πάρα πολύ που υποχρεώμαι ε, να το διαπιστώσω. Δεν είναι καθόλου καλό και για το κύριο και την εικόνα που δίνει το κοινοβούλιο. Αλλά ε, μια που μιλάμε για τους φόρους, δυστυχώς δεν ήταν εδώ ο Βολφ Κλίντς ε, όταν στην περασμένη έκθεση συζητήσαμε για τους φόρους και διαπληκτιστήκαμε και χρειάστηκε να μηνθώ εγώ, γιατί έχω μπουχτίσει για να το πω έτσι, συνεχώς να ε, παρουσιάζεται η χώρα μου ως δίθεν φορολογικός παράδεισος έχει πολύ μεγάλο δίκαιο όταν λέγει ο ίδιος ότι ο τρόπος με τον οποίο φορολογούν τα κράτη είναι ακόμα και παραμένει η δική τους κυριαρχή απόφαση. Και ξέρετε, δεν είμαστε μοσπονδιακό κράτος. Αν ήμασταν, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Ε, δυστυχώς δεν έχουμε φτάσει μέχρι και ορισμένοι ούτε να τα ακούσουν. Τότε θα μπορούσαμε να κάνουμε τέτοιες τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή και με χαρά να τις εγκρίνουμε γιατί δεν θα τις χρειαζόμασταν τότε, θα είχε λυθεί το θέμα. Αλλά τι να κάνουμε, δεν είμαστε ομοσπονδιακό κράτος, οπότε πώς έχουν τα πράγματα. Τα κράτη αποφασίζουν για τη φορολογία τους. Πώς ε, τα ρυθμίζουν αυτά. Εμείς στο Λουξεμβούργο είμαστε παράδεισος, μπορεί να είμαστε για το ΦΠΑ. Υπέρ των καταναλωτών είναι ο παράδεισος, καταναλωτικός παράδεισος και υπέρ εκείνων που κερδίζουν λιγότερα. Γιατί η καλύτερη κοινωνική πολιτική είναι χαμηλή έμεση φόρη. Χαμηλό ΦΠΑ. Στο Λουξεμβούργο είναι μεγαλύτερη η αγοραστική δύναμη όταν είναι 3% το ΦΠΑ ή 6-15% στα καταναλωτικά προϊόντα και στα τρόφιμα. Από ότι στη Δανία που έχουν φόρους στις μπανάνες, ξέρω εγώ, ε, ε, και στην Τζάγκουαρ 25% το ίδιο ΦΠΑ. Και χώρες που το κάνουν αυτό, που έχουν υψηλότερους άμεσους φόρους, δεν θα πρέπει να τους κατηγορούμε ότι είναι φορολογική παράδειση. Μα, ε, καλό είναι και χαίρομαι να λέτε ότι είμαστε φορολογικός παράδεισος για τους καταναλωτές και να παραμείνει. Παρένθεση ήταν όλο αυτό και πάω παρακάτω. Συμφωνώ βεβαίως απολύτως με τα όσα λέγει ο εισηγητής μας και οι σκιώδες. Αλλά συμφωνώ πολύ με τον εισηγητή ότι θα πρέπει το φορολογικό πλαίσιο να είναι ε, σταθερό, διαφανές και ε, αξιόπιστο. Ε, συμφωνώ απολύτως. Είμαστε κατά της διπλής φορολόγησης και κατά της διπλής αποφυγής φορολόγησης. Και είναι πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε και άλλη παρένθεση, Υπάρχει ένα τέτοιο θέμα στις χώρες όπου έχουμε ανταλλαγή πληροφοριών ε, για τη φορολόγηση των επιτοκίων. Διότι οι διάφορες διοικήσεις και έχουν έρθει και σε μένα υπάλληλοι και μου έχουν πει τι ωραία που είναι. Εγώ μένω στην Αγγλία, έχω και κάτι λεφτάκια στη Γερμανία και πουθενά δεν φορολογούμε γιατί οι διοικήσεις που ανταλλάσσουν εκατομμύρια πληροφοριών δεν μπορούν να τις επεξεργαστούν. Στις χώρες όμως που δεν υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών και δεν υπάρχει φορολόγηση και που πάντα παρουσιάζονται ως φορολογική παράθεση, τουλάχιστον πληρώνονται εκεί, καταβάλλονται οι φόροι από όλους στην πηγή. Πράγμα που δεν ισχύει στις χώρες που υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών γιατί δεν μπορούν να τις επεξεργαστούν και να τα εισπράξουν. Κλείνει και αυτή η παρένθεση. Συμφωνώ απολύτω λοιπόν με τον Βολφ Κλίντς ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει και διπλή και αποφυγή φορολόγησης από δύο χώρες, δηλαδή να μην φορολογείται κανείς πουθενά. Είναι περίπλοκα αυτά τα θέματα, αυτά ήθελα να πω και ζητώ συγγνώμη, Βολφ, για τα γερμανικούλια μου, αλλά ήθελα να τα πω στη γλώσσα σου. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Θα πρέπει να παραμείνουμε λογικοί και αυτές τις τρελές τροπολογίες που έχεις λάβει να τις απορρίψουμε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να κάνω ορισμένα σχόλια σε σχέση με τις τροπολογίες Νομίζω ότι πολλές φορές τονίσαμε ιδιαίτερα αυτούς τους ε, τελευταίους μήνες στην Επιτροπή. Μιλήσαμε για την, ε, σημασία της ανάπτυξης και του ανταγωνισμού. Γι' αυτό θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι ο κατακαιρματισμός των ε, χρηματοοικονομικών αγορών πλήττει την αγορά και το ε, κόστος χρηματοδότησης ε, των ΜΜΕ. Και ε, δεν χρηματοδοτούνται με βάση την οικονομική τους κατάσταση, αλλά με το που βρίσκονται. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο, μεγάλο λάθος και άδικο. η ΜΜΕ της ε, ευρωζώνης και του Ευρωπαϊκού χώρου δεν θα πρέπει να μην χρηματοδοτούνται κατά παρόμοιο τρόπο. Θα πρέπει να υπάρχει ε, ίση πρόσβαση στη χρηματοδότηση από τις ΜΜΕ. Γνωρίζουμε ότι αυτό πλήττει και την ανάκαμψη ορισμένων χώρων, όπως τη δική μου χώρα που έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια μεταρρύθμισης αλλά δεν μπορεί να ε, λάβει το αντίτιμο για αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια. Γι' αυτό θα πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι και οι ε, εθνικές τράπεζες και ε, γενικότερα όλοι οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Θα ήθελα να τονίσω ότι ο κύριος Κλίντς ε, προέβαλε μια πολύ καλή εργασία και θα ήθελα να του πω ότι χαίρομαι διότι λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη της ΜΜΕ που θα είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της οικονομικής ανάκαμψης. Δίνω ξανά το λόγο στον κύριο Κλίντς για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Δεν έχω να πω πολλά. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους. Και όπως είχα πει και εισαγωγικά, στην έκθεση αυτή εγώ δεν βλέπω να έχουμε θεμελιώδεις διαφορές και πέρα από κομματικά όρια των πολιτικών ομάδων και με αισιοδοξία ταινίζω την επόμενη εβδομάδα που θα συνεδριάσουμε στο Στρασβούργο και βάσει των συμβαστικών προτάσεων που θέλουμε να καταθέσουμε νομίζω μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα για την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Κλίντς. Θυμίζω ότι στην Επιτροπή μας θα ψηφίσουμε στις 22 Ιανουαρίου, ενώ στην Ολομέλεια θα πάει στη δεύτερη σύνοδο του μηνός Φεβρουαρίου. Λοιπόν, το σημείο 10 είναι διάφορα, δεν έχουμε κανένα διάφορο. Στις 11 ξέρετε ότι έχουμε μια κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Ελευθεριών. 15 λεπτά διάλειμμα.